Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε Πίμπαλξ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Διακοινοβουλευτική συνέδρο με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αναπτυξιακή πολιτική. Πριν ε, συνεχίσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποιες πληροφορίες. Έχετε ε, αυτά τα μπλε έντυπα. η Επιτροπή μας δεν έχει τη συνήθεια να χρησιμοποιεί αυτά τα έντυπα μπλε χρώματος. Αυτά ε, σας χρησιμεύουν για να εγγραφείτε να ζητήσετε το λόγο. Θα κάνουμε το εξής. Εάν ζητήσετε το λόγο, ε, το, ε, για αυτή τη στιγμή σηκώνετε το χέρι σας. Αν έχετε δώσει το μπλε θα μας δώσετε το μπλε είναι πολύ επίσημο αυτό το έγγραφο, αλλά εμείς το αγνοούσαμε, γι' αυτό θα προτιμούσα ε, να κάνουμε ό,τι κάνουμε συνήθως. Ε, είναι πολύ περίπλοκο να μάθουμε ε, και να κάτσουμε ένα τέταρτο να μάθουμε πώς λειτουργεί αυτό το play έντυπο. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε να λάβετε το λόγο, σηκώστε το χέρι σας ή αν θέλετε χρησιμοποιήστε το έντυπο. Είμαι η πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή για μένα να προεδρεύω αυτή τη ε, συνεδρίαση μαζί με τη συνάδελφο Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ, η οποία θα αναλάβει την προεδρία για το δεύτερο τμήμα της συνεδρίας. Η Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να καλωσορίσω τις αντιπροσωπείες των Εθνικών Κοινοβουλίων που είναι παρούσες εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση και ελπίζω η σημερινή συζήτηση να μας επιτρέψει να γνωρίσουμε αλλήλους λίγο καλύτερα, να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων μας και ή δυνατόν να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες διαβουλεύσεις και συνοχή ε, μεταξύ των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκών πολιτικών ε, της αρμοδιότητάς μας. Όπως προβλέπετε στην ημερήσια διάταξη, η συνεδρίαση θα γίνει σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα ε, μας ενδιαφέρει για να δούμε αν μπορούμε να πούμε ότι η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά εμπόδιο για τη μείωση της φτώχειας, ενώ στο δεύτερο τμήμα τίθεται το ερώτημα αν είναι εφικτή η τήρηση της ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα περιβάλλον με πληθώρα δωρητών. Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με κάποια συμπεράσματα για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για τη θέσπιση και τον έλεγχο της ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχάς όμως επιτρέψτε με να καλυσερώσω τον Άντρης Πίμπαλξ, όπως έκανα και προηγουμένως, είναι ο Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης. Ο κύριος Πίμπαλξ θα παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στη σημερινή συνεδρίαση. Κύριε Πίμπαλξ, έχετε το λόγο. Ah, merci, Madame la uh, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίε και κύριοι, πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία το να οργανώσει την ε, διακοινοβουλευτική συνάντηση ε, για αυτό το τόσο κρίσιμο θέμα για τα επόμενα έτη. Ξεκινώντα λοιπόν ε, θα ήθελα να παραθέσω από την έκθεση των ε, Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ελευθερία που αναφέρει η ανθρωπότητα δεν θα μπορεί να απολαύσει ασφάλεια χωρίς την ανάπτυξη. Δεν θα μπορεί να απολαύσει ανάπτυξη χωρίς την ασφάλεια. Και δεν θα μπορεί να έχει οράματα χωρίς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή πολιτική χωρίς ασφάλεια, καμία ε, πολιτική ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη και κανένα από αυτά ε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν είναι βαθιά ριζωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην προσέγγιση μας ε, στην ανάπτυξη. Έχει φτάσει λοιπόν η χρονική στιγμή ε, να δώσουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα τη θέση που τους αξίζει στην αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτό πρόκειται να κάνουμε με το όραμα το όραμα που έχουμε ένα έγγραφο στο οποίο προβλέπεται μια αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε. Το όραμα βασίζεται σε περισσότερο στρατηγική προσέγγιση για να ε, εξαλειφθούν ε, τα δεινά και απαιτείται να υπάρχει καλύτερη εστίαση σε καλή διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα, καλή και πιο σωστή εστίαση ε, στην επιδίωξη της αηφόρου ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες στόχος είναι και οι πόροι. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διοχετεύονται εκεί που χρειάζονται περισσότερο από όλα και εκεί που μπορούν πραγματικά να επιφέρουν αλλαγή. Και ποιος μπορεί να καταλάβει καλύτερα και να ενστερνιστεί αυτό το όραμα, γιατί θα πρέπει να το ξέρουμε η δική σας εμπειρία ε, στην ε, δημοκρατία ε, είναι μοναδική. Δεν είναι ένα ρομαντικό όραμα της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Πρόκειται για την ανάπτυξη ευφυών προϋποθέσεων. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε πολλά από τη Βόρεια Αφρική, τα ανθρωπινά δικαιώματα και η καλή διακυβέρνηση θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προσφέρεται η βοήθεια. Η αραβική άνοιξη έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο. Στον αραβικό κόσμο ε, οι νέοι έχουν πολύ μεγάλο θάρρος. Ε, ποιο είναι όμως το ρεαλιστικό κοινομάθημα που μπορούμε να μάθουμε από την αραβική άνοιξη. Μπορούμε να μάθουμε ότι τα παλιά ε, πρότυπα είναι πλέον πεπερασμένα. Πριν λοιπόν προχωρήσω θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, όσον αφορά ε, της, ε, την αιρεσιμότητα. Η αιρεσιμότητα δεν είναι προϋπόθεση για την περικοπή των κονδυλίων. η χρηματοδότηση καθορίζεται με βάση τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και την απόδοση της χώρας εταίρο. Μεγαλύτερη σημασία πρέπει να αποδώσουμε ε, σε, στην κατάσταση που αφορά στις χώρες σχετικά με την οικονομική τους διακυβέρνηση και γενικότερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι τα μαθήματα που μπορούμε να δώσουμε. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η αλληλεπίδραση πάνω σε οικουμενικές και συμφωνημένες αξίες. Τρίτον, ε, τα αποτελέσματα χρειάζονται χρόνο. Πολύ συχνά υπερτιμούμε αυτά που μπορούν να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα, όμως συστηματικά υποτιμούμε αυτά που μπορούν να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θα παραμείνει αδιάφορη στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να έχουμε ισορροπία ανάμεσα στα προληπτικά ε, και τα ε, μέτρα και τα μέτρα αντίδρασης. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σήμερα θα αναφέρω τέσσερα καθοριστικά στοιχεία. Πρώτον, πολιτικό διάλογο. Δεύτερον, ε, οικονομική συνεργασία για να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, περιοριστικά μέτρα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε ένα τέταρτο σημαντικό στοιχείο που είναι η συνέπεια στις πράξεις μας. Όσον αφορά λοιπόν την πρώτη διάσταση, το πρώτο στοιχείο του θέματος, ο πολιτικός μας διάλογος με τις γειτονικέ χώρες είναι καθοριστική σημασίας για να διασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, την καλλική διακυβέρνηση, ότι όλα αυτά αντιμετωπίζονται σε επίπεδο χώρας. Ο πολιτικός μας διάλογος βασίζεται ε, στον διαθρωμένο διάλογο, ε, σε συμφωνίες, σε συμφωνίες ad hoc και σε διαβουλεύσεις. Μέσα από αυτόν τον διάλογο ή αυτούς τους διαλόγους μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα σε ε, πρόορη φάση, αρκετά νωρίς. Αλλά ο διάλογος ε, πρέπει να είναι τακτικός, συστηματικός και να περιλαμβάνει την κοινωνία των πολιτών. Τέτοιου είδου δεσμεύσει αναφέρονται στο πρόγραμμα δράση για την ισότητα των δύο φύλων που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010. Και με βάση όλα αυτά ο διάλογο κατά κατώ τουλάχιστον με τις γειτονικέ χώρε θα περιλαμβάνει τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Οικονομικά και άλλα μέτρα ως αντίδραση στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μένει το τελικό καταφύγιο. <clears throat> Δεν πρέπει να υπάρχει μια στάνταρτ πρακτική. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μέτρα αυτά καθίστανται απαραίτητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, οι επιπτώσεις ε, περιοριστικών μέτρων πρέπει πάντα να λαμβάνονται πλήρως υπόψη. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα του τι ακριβώς ε, εννοώ τα ανθρώπινα δικαιώματα Συμπάμπου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα σχολιάσουμε. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να διακόψει τη βοήθεια προς την ε, Ζιμπάμπου εξαιρουμένη της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτή η αναστολή παρατάθηκε καθότι οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί δεν πληρώθηκαν. Αυτό δεν ήταν απόφαση κατά του λαού της Ζιμπάμπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί ή αναπτύσσει ανθρωπιστικές δραστηριότητες και συνεχίζει να στηρίζει προγράμματα που προσφέρουν άμεση βοήθεια στους ε, πολίτες. Ε, βοήθεια επίσης ε, και σε φορείς υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού. Έτσι λοιπόν τα περιοριστικά μέτρα δεν πρέπει να υπονομεύουν την υποστήριξη επιτόπου στους ανθρώπους. Και φτάνουμε στο τρίτο βασικό στοιχείο τη βοήθεια που παρέχουμε. Όλα τα εργαλεία της συνεργασίας ε, στηρίζουν τις ε, διαρθρωτικές ε, αλλαγές και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Προσφέρεται λοιπόν υποστήριξη συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης της δημιουργίας θεσμών, εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Έχουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για περιπτώσεις που κρίνονται ιδιαίτερα ευαίσθητες ε, και για χώρες όπου δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος ε, για την παρέμβαση κρατικών φορέων. Τα ευρωπαϊκά εργαλεία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν όπου η συνεργασία, αναστέλλεται η συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς. Υπάρχουν ε, θεμελιώδη θεμελιώδεις αρχές, με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δημοκρατικές ε, διαδικασίες. Κάθε εβδομάδα εμείς ε, προστατεύουμε τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τον τρόπο αυτό κάθε εβδομάδα ε, κατορθώνουμε να αποκαταστήσουμε θύματα κατάχρησης μεμονωμένα άτομα που πλέον δεν αντιμετωπίζουν κινδύνους. Ε, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτές μας τις προσπάθειες και είμαι σίγουρος αυτό ισχύει και για εσάς. Δεν αρκεί βέβαια αυτό. Μπορούμε να επιτύχουμε και πολλά άλλα. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τις ισχύουσες πρακτικές. Ε, μπορούμε να επηρεάσουμε το δημοκρατικό μέλλον των ε, εταίρων μας. Από προσωπική εμπειρία γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει να ζει κανείς σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι εγώ θα ανεχτώ η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η βοήθειά της ε, να δίδεται υπό αμφισβήτηση ή αν δεν πρέπει να δοθεί, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Γι' αυτό και θα υπάρξει αναθεώρηση των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Έτσι λοιπόν έχουμε μία μοναδική ευκαιρία για να συμπεριληφθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα περισσότερο στις ε, πολιτικές που εφαρμόζουμε. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να στρέφουμε το βλέμμα πέρα από τα ε, απλά εργαλεία. η υποστήριξη του, ε, η δημοσιονομική υποστήριξη είναι μια πολύ καλή προσέγγιση. Μια προσέγγιση που μας επιτρέπει να επιτύχουμε, να επιδιώξουμε βασικούς στόχους ε, με χώρες εταίρους, ενώ παράλληλα εμπλεκόμεθα και σε διάλογο με την κάθε κυβέρνηση, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη κυρίως όταν αναλύουμε το προφίλ μιας χώρας. Ε, και από εκεί κρίνεται και κατά πόσο αξίζει τον κόπο να τη στηρίξουμε οικονομικά. Αυτές λοιπόν οι τρεις διαστάσεις, αυτά τα τρία στοιχεία καθορίζουν τον δρόμο. Ε, βέβαια ε, αυτό που είναι καθοριστικό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια ανάμεσα στον πολιτικό διάλογο και τα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση που την ανέφερα, σας είπα προηγουμένως, είναι η συνέπεια στις πράξεις μας. Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συμβούν όλα αυτά. Εδώ έχουμε έναν κατάλογο με στοιχεία, δηλαδή πρώτον, πρέπει να προαχθεί περαιτέρω μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά στην συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα διάφορα κοινοτικά εργαλεία. Αυτό να εφαρμόζεται συστηματικά, ξεκινώντας με τη φάση του σχεδιασμού. Δεύτερον, η οικονομική διακυβέρνηση και οι στρατηγικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να προετοιμάζονται από τις αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με τα κράτη-μέλη και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια συγκεκριμένη χώρα. Βοηθούν όλα αυτά ε, στο να επιτυγχάνεται μεγαλύτερο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρίτον, τα ανθρώπινα δικαιώματα εμφασίζονται και στην μέση διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό πρέπει να συμβαίνει και σε άλλου διεθνείς οργανισμούς και σημαντικά δωρητές. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, σημαντικός διεθνής παίκτη και μπορεί κατόπιν τούτου να ε, στρέψει περισσότερο την προσοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη αλλά και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργούν περισσότερο προληπτικά, θα σκούν εκ των προτέρων πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγαπητά μέλη, δεν μου αρέσει η λέξη αιρεσιμότητα. Ο στόχος μας είναι να στηρίζουμε ε, τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, αλλά για να είναι η όλη διαδικασία βιώσιμη είναι απολύτως απαραίτητο τα ανθρώπινα δικαιώματα να παραμείνουν υψηλά στην ε, ημερήσια διάταξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίμπαλξ. Σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Επίτροπε και τον κύριο Φερνάντες για την παρουσίαση τους εδώ και για το γεγονός ότι παρουσίασαν την άποψη των θεσμικών τους οργάνων για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Φερνάντε ο οποίος θα μας παρουσιάσει την άποψη της, εξωτερικής υπηρεσίας, ε, της υπηρεσίας εξωτερική δράσης. Κύριε Φερνάντε, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ εκ μέρους της, είπα, της εκπροσώπου, της Βαρόνης Άστον, για να παρουσιάσω την άποψη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Βεβαίως το να λαμβάνει κάποιος το λόγο μετά από τον Επίτροπο είναι δύσκολο πάντα, διότι πολύ εύγλωτα παρουσίασε πολλά από τα στοιχεία τα οποία ήθελα να σας παρουσιάσω κι εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποια σημεία από αυτά τα οποία ανέφερε, ιδίω στη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί πρέπει να δούμε και την αναπτυξιακή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ασφάλεια από κοινού, αλλιώς δεν θα υλοποιηθούν. Επίσης να σας πω ότι ο τίτλος της σημερινής συζήτησης υποδηλώνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναπτυξιακή πολιτική φαίνεται να πηγαίνουν η μία αντίθετα στην άλλη και δεν ξέρω εάν ε, είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι εργάζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθούμε να προωθήσουμε και την ανάπτυξη. Και αυτό λέει και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και η συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και συμπεριλαμβάνει και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αναπτυξιακή πολιτική. Άρα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι. Και νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεκινούμε υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι δύο πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω και το θέμα της εφιούς αιρεσιμότητας που ανέφερε ο Επίτροπος. Ε, έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τον πολιτικό διάλογο, πολλά να κερδίσουμε από τη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να άρουμε και τους φραγμούς και την, ε, ε, να διασκεδάσουμε την αντίληψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αιρεσιμότητα μπορεί να έχουν αρνητική επίπτωση για την αναπτυξιακή πολιτική. Δεν θα πρέπει να το πιστέψουμε κάτι τέτοιο, γιατί εμείς στην Ευρώπη προσπαθούμε να προχωρήσουμε προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση, ότι το ένα προωθεί το άλλο, συνεργάζονται μεταξύ των και πηγαίνουν χέρι-χέρι, όπως είπε και ο Επίτροπος. Δεύτερο, η συνοχή και το συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε να προσπαθήσουμε οι εξωτερικές μας δράσεις, οι δράσεις εξωτερικής πολιτικής, ε, οι ε, δράσεις ανάπτυξης να είναι συνεκτικές και να προσπαθούν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο. Είτε είναι στόχοι για τη μείωση της ένδυας, είτε είναι στόχοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί θα πρέπει όλα να εξετάζονται από κοινού και να έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο. Προωθούμε ήδη 40 διαφορετικούς διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Προχωρούμε κάποιες στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες σχεδόν τις τρίτες χώρες του κόσμου. Και φυσικά ετοιμαζόμαστε για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που μόλις σας εξήγησε ο Επίτροπος. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική η στιγμή αυτή, διότι θα προσπαθήσουμε να δούμε το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, τη συνοχή και την εξωτερική μας δράση. Η υπηρεσία μας μαζί με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τη σκέπη του Επιτρόπου Πίμπαλξ και της ε, Κάθριν Άστον θα μπορέσουν να διαδραματίσουν σημαντικά ρόλο και νομίζω ότι αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες προτεραιότητες ώστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναπτυξιακή πολιτική να εργαστούν συνεκτικά. Ο κύριος Πιμπάλ ξαναφέρθηκε προηγουμένως στον πολιτικό διάλογο. Θεωρώ ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα διπλωματικό εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σθένος προκειμένου να γίνουν προτεραιότητα η αναπτυξιακή πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της φιούς ερεσιμότητας, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και αυτό βάσει των τεσσάρων κριτηρίων που αναφέρατε και θα πρέπει να αναφέρω και ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο νομίζω ότι θα συζητηθεί και αργότερα σήμερα το απόγευμα. Εξ όσων κατανοώ και χαίρομαι γι' αυτό έχουμε εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ. Έχουμε ένα νέο κόσμο λοιπόν με νέους δωρητές και νέους παράγοντες και αυτή η συνοχή και αυτό το συνολικό στοιχείο θα πρέπει να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία μας για κοινό προγραμματισμό, για το πώς μπορούμε να έχουμε κοινέ προσεγγίσεις με τα κράτη-μέλη σε τρίτες χώρες, με νέους δωρητές και με τους νέους παράγοντες που αναδύονται και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανασκουμποθεί όσο μεγαλύτερη βαρύτητα μπορέσει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο καλύτερα θα διαβιβάσουμε το μήνυμά μα. Το μήνυμά μα είναι σαφέ για την ανάπτυξη, το μήνυμά μα είναι σαφέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να του προσδώσουμε και τη δέουσα βαρύτητα. Και νομίζω ότι εδώ τα Εθνικά Κοινοβούλια και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να αποστείλουν τα σωστά μηνύματα, τα οποία νομίζω ότι πρέπει να αποστείλουμε άλλοι ε, με τη δέουσα βαρύτητα, όπως είπα προηγουμένως, ώστε να έχουν αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό, να διέπεται το μήνυμά μας από την κατάλληλη βαρύτητα για να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι προωθούμε επίσης ε, αντίστοιχες συνεδριάσεις και χαίρομαι για το γεγονός ότι ε, συνεδριάζουν ε, οι συνεδριάσεις αυτές εδώ, γίνονται οι συνεδριάσεις αυτές εδώ για, με κοινέ επιτροπές και θα πρέπει να προσπαθούν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή Ανάπτυξης να εξετάζουν τα θέματα αυτά από το κοινό οπτικό πρίσμα που θα έπρεπε να τις διέπει. Και με αυτό νομίζω θα ήθελα να ολοκληρώσω, να σας ευχαριστήσω διότι προσκαλέσατε την ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε εδώ με ποιο τρόπο μπορεί να συνεισφέρει και η υπηρεσία μας και ε, να σας υπενθυμίσουμε ότι αποτελούν και βασική μας προτεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανάπτυξη και μάλιστα από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τον Επίτροπο και τον κύριο Φερνάντε Σό για την παρουσία τους εδώ σήμερα στην ε, συνεδρίασή μας και για το γεγονός ότι μας παρουσίασαν την άποψη των θεσμικών τους οργάνων για τη συγκεκριμένη συζήτηση. Μετά λοιπόν από αυτή την εισαγωγή των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Περνάμε στο πρώτο τμήμα της συνεδρίασης. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα του κατά πόσον μπορούμε να πούμε ότι η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά εμπόδιο για τη μείωση της φτώχειας. Τα θέματα της ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν είναι αλληλένδετα. Θεωρούμε ότι υπάρχει όλο και περισσότερη συνένεση για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσέγγιση στην οποία όχι μόνο ε, τα αστικά και ε, πολιτικά δικαιώματα αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα να ε, θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και η συνεργασία με τα τρίτα κράτη που προβλέπουν και χρηματοοικονομική βοήθεια πρέπει να απαιτεί ίσως να υπάρχει και σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ορισμένες φορές έχουμε αναστολή της βοήθειας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε καταστρεπτικές συνέπειες, κυρίως για θέματα ένδυας. Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι αυτές που πλήττονται, χωρίς να πλήττονται οι ελίτ και οι πλουσιότεροι. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πιο ευφυείς κυρώσεις, ε, οι οποίες θα πρέπει να κερδίσουν έδαφος. Και αυτές φυσικά θα πρέπει να στρέφονται σε οικονομικές και πολιτικές ελίτ ή σε συγκεκριμένους ε, τομείς ε, της ε, ε, κοινωνίας που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τη σημερινή συζήτηση. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε και κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε βοήθεια στις πιο ευάλωτες πτυχές των πιο στερημένων χωρών, όπου έχουμε και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τι γίνεται όταν δεν υπάρχει συνεργασία με ε, βασικές οργανώσεις ή κατά πόσον θα έπρεπε να ε, μην υπάρξει πια αυτή η ρήτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή να επικεντρωθούμε ίσως στα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Θα μπορούσαμε ίσως να συνδυάσουμε και μια ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κάποια ενθαρρυντικά βήματα ή σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια νεοτροπία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βοηθήσουμε ταυτόχρονα την ανάπτυξη των χωρών αυτών. Επειδή λοιπόν έχουμε και εκπροσώπους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια εδώ, θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε και ποιοι παράγοντες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα για το πώς θα εφαρμόσουμε τα μέτρα, πώς θα υποπτεύσουμε στη συνέχεια και θα αξιολογήσουμε ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε συμφωνίες συνεργασίες και στο διάλογο για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε συνεκτική εφαρμογή και σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο και να συμπεριλαμβάνεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ε, συνέχιση ή την αναστολή της αναπτυξιακής βοήθειας ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Να δώσουμε λοιπόν και στους ευρωβουλευτές και στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν ζητήσει το λόγο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με δύο εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και επειδή είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να παρέμβουν, το πολύ πέντε λεπτά σας παρακαλώ κάθε ομιλητής θα σας διακόπτω στα 5 λεπτά. Αρκετό είναι ο χρόνος, ούτως ή άλλως λιγότερο δίνουμε συνήθως. Στα 5 λεπτά θα σας διακόπτω είτε έχετε ολοκληρώσει είτε όχι, αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Η κυρία Γκρέζ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εργανώστε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση και θα ήθελα να επισημάνω την ευθύνη των κοινοβουλίων σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Υπάρχει νομοθεσία, διότι σε όλες τις συμφωνίες υπάρχει μια ρήτρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο Επίτροπος προηγουμένως έχθε το δάκτυλο από τον τύπο των ήλων, εξηγώντα ότι πολλές φορές είναι ο πληθυσμό αυτός ο οποίος πλήττεται και υπόκειται τις συνέπειες. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να σταθώ σε αρκετές ε, πτυχές. Οι ρήτρε αυτές νομίζω ότι δεν επαρκούν. Είναι απαραίτητες αλλά δεν επαρκούν. Υπάρχει ανάγκη μαζί ε, με τους σαφείς μηχανισμούς ε, να δίνεται και η βοήθεια και ταυτόχρονα να υπάρχουν και διαδικασίες διαβουλεύσεων των ενδιαφερομένων. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε από τα έξω το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σταθώ σε κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ αλλά νομίζω ότι αρμόζει να συζητηθεί. Είναι το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων που είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώνω ότι υπάρχουν ε, αρκετά μέτρα. Υπάρχουν αφενός εμπορικοί κανόνες οι οποίοι είναι πολύ δεσμευτικοί. Ο Επίτροπος Εμπορίου, εξ όσων μαθαίνω, θέλει να αποκλείσει την πρόσβαση στις αγορές για όσους δεν έχουν υπογράψει τις ανάλογες συνθήκες. Και επίσης υπάρχει και η κοινωνική βοήθεια. Άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περάσει στα θέματα του ΠΟΕ την ανάγκη της ρήτρα κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεύτερον, και υπενθυμίζω ότι είχα παρουσιάσει και μία έκθεση ε, για γνωμοδότηση η οποία είχε ψηφιστεί για θέματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά παρόλα αυτά η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι μόνο επιθελούσια βάσεω ακόμα. Και τρίτον, το θέμα των κυρώσεων, χωρίς καμία παρακολούθηση στη συνέχεια για το κατά πόσον εφαρμόζονται οι κανόνες ε, για τις συμφωνίες αυτές. Προς τον Επίτροπο λοιπόν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Πώς θα μπορέσετε να υλοποιήσετε δεσμευτικούς κοινωνικούς κανόνες που να αφορούν και την, ε, ε, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς θα μπορέσετε να φροντίσετε να υλοποιηθούν οι κανόνες των συμβάσεων και να ε, εφαρμοστούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάμνουρ έχει το λόγο. Δεν ξέρω αν είπα σωστά το όνομά σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η επικέντρωση της πολιτικής σε τέτοια θέματα αποτελεί μία συνέπεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1948 από την Ηνωμένα Έθνη αποτέλεσε το μοναδικό εργαλείο για την συμφιλίωση της ανθρωπότητας μετά από την τεράστια αυτή σύγκρουση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να επενέσουμε τους πολιτικούς της εποχής εκείνης για το γεγονός αυτό. Γιατί στις χώρες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν σωστά και καλά ανεπτυγμένα τότε. Δυστυχώς τα ανθρώπινα, τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι υποχρεωτικά. Δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσον η σημερινή νομοθεσία βοηθάει όντω τα ανθρώπινα δικαιώματα ή όχι. Είναι σημαντικό να βρεθούν νέες πολιτικές οι οποίες θα δώσουν απαραίτητες εγγύησεις για τα ατομικά δικαιώματα και αυτό αφορά και τις εθνικές πολιτικές αλλά και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, το εσωτερικό της κοινωνικής πολιτικής. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε τη φτώχεια στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη τέτοιων πολιτικών που ως σκοπό θα έχουν την καταπολέμηση της ένδυας πάντα θα πρέπει να συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. μια αξιοπρεπή ζωή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Η κοινωνική ανισότητα βρίσκεται στον πυρήνα των συγκρούσεων σε όλον τον κόσμο. Και αυτό γιατί ο κόσμος δεν έχει τα μέσα για να πετύχει αυτά που χρειάζεται στην αγορά εργασίας και η βοήθεια θα πρέπει να ε, διανέμεται με καλύτερο τρόπο, γιατί η φτώχεια είναι κακός σύμβουλος. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, συνήθω υπάρχει ένα μικρό κενό για να ακούω και την ε, μετάφραση. Ο λόγος στον κύριο Κάσμαν, πέντε λεπτά το πολύ, έτσι, αν... Ε, ε και τρία λεπτά ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλώ ως ηγητής της αναθεωρημένης Συμφωνίας Κοτονού είναι ενδιαφέρον που και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και από τον Επίτροπο ακούσαμε την ε, παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω ε, και να θέσω κάποια σχόλια. Αν η αιρεσιμότητα αποτελεί αρνητικό στοιχείο σε ό,τι αφορά την μείωση της φτώχειας, πώς θα διασφαλίσουμε ότι πληρούνται όντως και τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να κοιτάξουμε τις, χώρες, με τις οποίες έχουμε τις συμφωνίες, τη Συμφωνία Κοτονού. Υπάρχει άρνηση από τις χώρες αυτές επί της τροποποιημένης ρήτρας. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα θέματα μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει σεξουαλικής προτίμησης από τις 49 από τις 79 χώρες ΑΚΕ υπάρχει ποινική δίωξη της ε, ομοφιλοφιλίας μέχρι ε, και φυλάκισης στην Αφρική 38 χώρες ε, θεωρούν ποινικό αδικήμα την ομοφιλοφιλία. Τι πετύχαμε λοιπόν με το διάλογο αυτό, τι πετύχαμε με, με την μεικτή διακοινοβουλευτική ομάδα. Τα μέλη των χωρών ΑΚΕ εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και το ενδεχόμενο συζήτηση Άρα έχουμε συμφωνίες όπως το κοτονού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόσαμε τις ρήτρε αναστολής ή κυρώσεων βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν το δυναμικό μας, αλλά στις χώρες αυτές έχουμε οργανώσεις που κάποιες φορές μιλούν για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων για τα δικαιώματα των σεξουαλικών μειονοτήτων. Αλλά διώκονται αυτές οι οργανώσεις και τελικά κλείνουν. Ερωτώ λοιπόν και την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τι μπορούμε να κάνουμε όταν δεν μας ακούν και όταν η πίεση από τους ομοτήμους δεν λειτουργεί. Το Κοινοβούλιο κατά την επικύρωση της νέας αναθεωρημένης συμφωνίας νου, όταν ανακύπτουν ερωτήματα, τι θα κάνει, να σας πω ότι δεν πρόκειται για μια αστεία ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπε και ο προηγούμενος ε, ομιλητής, το θέμα είναι να βάλουμε το άτομο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Πολύ σωστά το είπε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αρχές τις οποίες υπονομεύουμε. Αν δεν έχουμε αξίες ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν εφαρμόζουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα καταλήξουμε να καταστούμε μια οικονομική κοινότητα και μάλιστα ε, που δεν λειτουργεί. Αν δεν έχουμε τίποτα παραπάνω... Κοιτάξτε, είμαστε μια οργάνωση που έχει ανθρώπινες αξίες και να κλείσω λέγοντας ότι αν οι χώρες ΑΚΕ δεν κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός, είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής τους. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με τους μεγάλους δωρητές για το θέμα αυτό, σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη και την Παλαιστίνη όπου τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία εδώ πέρα εμείς θεωρούμε αυτονόητα, δεν αναγνωρίζονται, όπου έχουμε, Ισρα... έχουμε συμφωνία εμπορικής σχέσης με το Ισραήλ και μόλις μία φορά έχει γίνει αίτηση για αναστολή της συμφωνίας αυτής και το Συμβούλιο αρνήθηκε. Τι μήνυμα άραγε αποστέλνουμε στον υπόλοιπο κόσμο όταν ζητάμε να μας παίρνουν στο σοβαρά και εμείς οι ίδιοι δεν εφαρμόζουμε τις ίδιες μας τις συμφωνίες σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κανονικών ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται ε, λόγω των, της προέλευσής τους, λόγω της διαφορετικότητάς τους. Είναι απαράδεκτο και θα ήθελα η Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να απαντήσουν τις ερωτήσεις μου χωρίς διάλογο. Τι μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Είχα ζητήσει και εγώ το λόγο και θα λάβω το λόγο, αλλά θα ήθελα απλώ να συνεχίσω αυτά που μόλις είπε ο κύριος Κάσμαν. Θα είμαι πιο σύντομη όμως, διότι τα ουσιώδη ε, έχουν ήδη λεχθεί και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Πίμπαλξ, ότι η αριθμότητα δεν αποτελεί πρόσκομα και δεν θα πρέπει να κάνουμε σύγχυση μεταξύ των ανθρωπιστικών θεμάτων και της ανάπτυξης, διότι τα ανθρωπιστικά ζητήματα ε, είναι ανθρωπιστική βοήθεια στους πιο ευάλωτες, ενώ η αιρεσιμότητα ποιου θα πλήξει. Θα πλήξει αυτούς οι οποίοι ε, είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό εάν πληχθούν οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι. Θα σταθώ στην Ουγκάντα. Όπως γνωρίζετε στην Ουγκάντα οι ομοφιλόφιλοι καταδικάζονται σε θάνατο. Εάν είστε γονείς ομοφιλόφιλου ε, καταδικάζεστε σε φυλάκιστη γιατί δεν μπορείτε να φτιάχνετε ομοφιλοφίλους. Έτσι λένε τα κείμενά τους εκεί. Αν είστε ιδιοκτήτης και νοικιάσετε ένα διαμέρισμα σε ομοφιλοφίλους καταδικάζεστε σε φυλάκιση σήμερα, τη σήμερον ημέρα, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να δίνεται βοήθεια σε χώρα αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ τη χώρα αυτή που έχει, τις χώρες, συγγνώμη, τη Γερμανία και δεν ξέρω και κάποιος άλλος, δεν τις γνωρίζω όλες τις χώρες που έχουν αρχίσει να μην βοηθούν. Είχα πάει στην Κινσάσα και πήγα και στο Κιβού οι γυναίκες βιάζονται ε, σε καθημερινή βάση ε, όπως πηγαίνει ε, κάποιος να αγοράσει ψωμί στο φούρνο. Μετά από τις τρεις μέρες λοιπόν που πέρασα στο Κιβού και πήγα στη συνεδρίαση των χωρών και στην Κινσάσα δεν άκουσα κουβέντα για αυτό το πράγμα. Ζήτησα το λόγο για να μιλήσω και σχεδόν μου είπαν οι επικεφαλείς των χωρών ΑΚΕ ότι ψεύδομαι, ενώ τα είδα. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ε, πήγα στο κυβού και τα είδα. Σήμερα γίνονται συνεχώς συνεθριάσεις στην περιοχή μου με ε, την κοινότητα των λεσβιών ομοφιλοφίλων ε, κλπ. και με αρκετούς ε, από αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να σας πω ότι οι Γάλλοι πολίτες και οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν αντέχουν άλλον αυτή την κατάσταση. Οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν πώς είναι δυνατόν, ενώ σήμερα βιώνουμε όλη την κρίση στις ευρωπαϊκές χώρες, κάποιες χώρες πλήττονται περισσότερο από κάποιες άλλες και οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται γιατί συνεχίζουμε να δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες ΑΚΕ, οι οποίες δεν σέβονται ούτε τα ελάχιστα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές είναι πρακτικές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και χρόνια, αλλά σήμερα πλέον τα πράγματα αλλάζουν, ο κόσμος αλλάζει. Οι πολίτες δεν είναι πλέον ακακαρνάκια που εμπιστεύονται τους πολιτικούς και όλους τους υπολείπους. Επομένως, ήγηκε η ώρα να πούμε φτάνει, δεν θα το δεχτούμε πλέον. Και πραγματικά εγώ θα ήθελα να σας ζητήσω θερμά να υποστηρίξετε την εφαρμογή αυτής της ρήτρα για τις χώρες που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα λέμε ότι πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για τα κριτήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα τελεία και παύλα. Οι χώρε ΑΚΕ είναι αυτέ οι οποίε πρέπει να μάθουν ποια είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πρέπει εμεί να προσαρμοστούμε εμεί στα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζουν οι διάφορε χώρε. Νομίζω ότι αυτό θέλετε να πείτε κι εσεί. Κύριοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, φτάνει. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει το λόγο η κυρία Μπέις. Ζητώ συγγνώμη για την προφορά του ονόματος, δεν σας γνωρίζω γι' αυτό. Από την Αυστρία. Μπέις, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Μπέιερ το όνομά μου. Ah, B-A-Y-Z. <laughs> <laughs> Δεν το έχω γραμμένο σωστά, θα μπορούσα να το είχα πει. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις ερωτήσεις που έτιαξαν. Καταρχήν δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το κατά πόσον ε, έχουμε κοινό ορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μένα είναι απόλυτα σαφές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, ισχύουν για όλους, ε, είναι συνεδεμένα με όλους τους πολίτες του κόσμου αλλά γνωρίζουμε ότι το σύνταγμα πολλών κρατών έχει τέτοια μορφή έτσι ώστε να μην προβλέπει τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Πολλές φορές συντάγματα δεν προβλέπουν διαχωρισμό εξουσιών, ε, δεν προβλέπεται νομική προστασία. Άρα δηλαδή, δείτε το ερώτημα, ε, πώς ακριβώς ε, ερμηνεύουμε όλοι μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν καν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πώς μπορούμε να καταλήξουμε λοιπόν σε μια κοινή ερμηνεία. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εξή. Στην περίπτωση των ε, προϋποθέσεων και των κυρώσεων, όταν οι παραβιάσεις ε, γίνονται από ανθρώπινες κυβερνήσεις, επιβάλλεται κύρωση να μην χορηγείται ανθρωπιστική βοήθεια και ανταυτού επιθυμούμε να στηρίξουμε την, την κοινωνία των πολιτών. Αλλά ποια κοινωνία των πολιτών. Μία κοινωνία των πολιτών η οποία αναγνωρίζει τα οικουμενικά, ανθρώπινα δικαιώματα ή μήπως υπάρχει και μια σκοτεινή πλευρά της ε, κοινωνίας των πολιτών και αν ναι Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Το τρίτο που δεν είναι σαφές στη συζήτηση είναι για ποια ανθρώπινα μιλάμε. Της πρώτης, της δεύτερης, ε, της ε, τρίτης γενιάς ή για όλα. Μιλάμε για τα αρχικά, αυτά που έχουν ε, εγκρίνει τα Ηνωμένα Έθνη. Μιλάμε για κοινωνικά, πολιτιστικά, μιλάμε για δικαιώματα που βασίζονται, δράζονται στο διεθνές δίκαιο. Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε τελικά. Θέλω επίσης να παρατηρήσω ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε πολιτικές της ε, δεν σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματο χάρη, η ευρωπαϊκή πολιτική πρώτων υλών, η πολιτική αυτή ε, δεν νομίζω ότι έχει κατά νου τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ή η πολιτικη αλίας, όπως χαράστε μέχρι τώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή έχει κλείσει και τα δύο μάτια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μένα αυτά είναι μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος Θέλω να, κάνω, να θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές εμπορικές συμφωνίες, ε, ε, συμφωνίες ε, προστασίας επενδύσεων που περιλαμβάνουν και ρήτρε σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δούμε όμως την ενέργεια που χρησιμοποιείται για να εφαρμοστούν, ελοποιηθούν οι οικονομικές ρήτρες και πόσο λίγη είναι η ενέργεια που χρησιμοποιείται για να εφαρμοστούν οι ρήτρε περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα δείτε ότι υπάρχει παντελής ανισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει τι είδου ερωτήσει μπορούμε να βρούμε όλοι από κοινού, έτσι ώστε αυτά που αναφέρονται στα χαρτιά να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κάσμαρεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Μου άρεσαν πολύ αυτά που είπε ο Επίτροπος Πίμπαλξ για την ε, αμοιβαιότητα στις σχέσεις που θα πρέπει να υπάρχει και αυτά που ακούσαμε και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Ράσης σε ό,τι αφορά τους ευφυείς όρους. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Όταν πρόκειται για κράτη τα οποία δεν ε, μοιράζονται τις ίδιες μου τις ίδιες ε, απόψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν ούτε ευφυείς όροι, ούτε διάδραση στην περίπτωση αυτή και νομίζω ότι έδωσαν και ο κύριος Κάσμαν και η συνάδελφος ε, καλά παραδείγματα. Στο Δεκέμβριο έχουν περάσει, έχουμε 10 χρόνια από τη φυλάκιση ενός ε, δημοσιογράφου στην Ερυθρέα ο οποίος είναι σουηδικής προέλευσης. Κάναμε συζητήσεις σχετικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ άλλων και με πρωτοβουλία του κυρίου Μπούζεκ ε, αναλάβαμε πρωτοβουλίες. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει φυλακιστεί εδώ και 10 χρόνια αν ζει καν. Παρά το γεγονός ότι έχει σουηδική υπηκότητα, επαναλαμβάνω. συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ και ρωτήσαμε ευθέως ε, τους εκπροσώπους της Ερυθρέας κατά πόσον ζει ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Ακούσαμε μία μακρά ομιλία για τα ανθρώπινα και δικαιώματα στην Ερυθρέα. Τυπικούρες ακούσαμε, αλλά δεν μας απάντησε ευθέως αν ο κύριος αυτός ακόμα βρίσκεται εν ζωή ή όχι. Ο συνάδελφος Όλης Σμίτ, ο οποίος ασχολείται με τα θέματα αυτά, εξανέστη, σηκώθηκε και οι συνάδελφοι από την Αφρική του επιτέθηκαν λεκτικά κατηγορώντας τον για αγένεια. Έμα ε, θα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής. Όταν δεν υπάρχουν κοινοί παρανομαστές, όταν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε βασικά ζητήματα, δεν μπορούμε σε επίπεδο εταιρικό, σε διακοινοβουλευτικές συνελεύσεις να συνεννοηθούμε. Αυτό τι σημαίνει ότι η Ερυθρέα δεν χρειάζεται τη συνεργασία μας. Όχι, τη χρειάζεται, αλλά μεγάλο τμήμα και του δικού μας προπολογισμού διατίθεται για το στρατό. Και αυτό χρηματοδοτεί ουσιαστικά την ενόπλη σύγκρουση με, τους, με τις γειτονικές ε, χώρες της Ερτρέας. Όλα αυτά λοιπόν μου φαίνονται ακραία. Θα πρέπει όμως να μπορούμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένες απαντήσεις ε, από την Ερυθρέα για το κατά πόσο ζει αυτό το άτομο ή όχι. Η οχι Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε να καλωσορίσω με τη σειρά μου τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και ιδιαίτερα κάποιους φίλους με τους οποίους κάνουμε αγώνα σε παγκόσμιο επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαίρομαι που τους βλέπω εδώ. Κυρία Πρόεδρε, η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συνώνυμη με τον εκδημοκρατισμό, με την δημοκρατική παιδεία και με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα τον Επίτροπο ε, ότι δεν θα ανεχθεί την παραχώρηση αναπτυξιακής βοήθειας σε μη δημοκρατικά σε δικτατορικά καθεστώτα που για μένα μεταφράζεται σαν δέσμευση ότι δεν θα παρατηρήσουμε ξανά το φαινόμενο να συνεργαζόμαστε για χρόνια με δικτατορικά, με στιγνά δικτατορικά καθεστώτα και στη συνέχεια όταν υπάρξει εξέγερση του λαού να θυμηθούμε και λίγο τον λαό, να πάμε να τον βοηθήσουμε. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο πράγμα η επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια για να βοηθήσουμε ένα πληθυσμό να επιβιώσει και άλλο είναι η αναπτυξιακή βοήθεια. Όσον αφορά την επίγουσα βοήθεια για να ζήσει ένα λαός, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε και πολύ υπόψη το επίπεδο της δημοκρατίας, γιατί πρέπει να ζήσουν, πρέπει να φάνε για να ζήσουν δεν πρέπει να αφήνουμε και την, την βοήθεια να πέφτει στα χέρια εκείνων που θα την πουλήσουν, θα την μοσχοβουλήσουν παραπέρα. Όσον αφορά όμω την αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να, να θυμόμαστε ότι οι δρόμοι που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι βασικά τρει. Είτε πρώτα θα περιμένουμε να υπάρξει εκδημοκρατισμό και στη συνέχεια να αρχίσει να παραχωρείται η αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το λέμε, αλλά δεν μπορεί να, να το εφαρμόσουμε στην πράξη είτε να δίνουμε την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά να λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος και το ρίσκο να ε, αναπτύσσεται παράλληλα και η διαφθορά, να ε, πέφτει η βοήθεια στα χέρια διεφθαρμένων καθεστώτων, είτε να παρατηρείται εκ παραλλήλου ανάπτυξη Ινστιτούτων Εκδημοκρατισμού και Δημοκρατικής Παιδείας με παράλληλη λειτουργία πυρήνων ε, ανάπτυξης στην κοινότητα με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτουμε την, τους διεφθαρμένες κυβερνήσεις και αυτό νομίζω ότι είναι ο πλέον επιτυχής τρόπος. Η ύπαρξη πολλών μεγάλων δωρητών, χωρί να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό αναπτυξιακό συντονιστικό κέντρο, εγκυμονεί τον κίνδυνο η βοήθεια να φτάνει σε διεφθαρμένου παράγοντε. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και γι' αυτό και το πρωί σήμερα μιλούσαμε προ αυτή την κατεύθυνση, για την λειτουργία αυτού του κέντρου. Ε, Θέλω να επιμείνω και σε μια άλλη βασική μου θέση, την οποία επαναλαμβάνω πάντοτε, ότι δεν μπορεί να δίνεται αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρε οι οποίε κινούνται συνεχώ προ την κατεύθυνση των εξοπλισμών ή παράγουν πυρηνικά, αν θέλετε να το πάμε παραπέρα, πυρηνικά όπλα. Και να σα θυμίσω το παράδειγμα τη Αιθιοπία, όπου για πάρα πολύ καιρό δουλεύαμε όλοι να στείλουμε αναπτυξιακή βοήθεια και την ίδια μέρα τα αιθιοπικά αεροπλάνα εμβομβάρδιζαν την Ασμάρα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τονίνη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με την ε, ρεαλιστική προσέγγιση του Επιτρόπου και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δηλαδή να έχουμε ευφυείς όρους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι εγώ θεωρώ ότι ο καλύτερος δυνατός τρόπος για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μέσω διαλόγου. Σε γενικές γραμμές, για λόγους αρχής, ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να γίνει μια συζήτηση ε, με μία χώρα εταίρο παρά ε, να σταματήσουν ε, οι σχέσεις μεταξύ μας. Ακόμα και αν είναι δύσκολη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να κάνω διάκριση μεταξύ δύο επιπέδων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφενός υπάρχει το πολύ περίπλοκο και αποφασιστική σημασία ζήτημα της μετάβασης προς τη δημοκρατία και εμείς γνωρίζουμε ότι ο εκδημοκρατισμός ε, σε πολλές χώρες είναι μια μακρά διαδικασία η οποία απαιτεί υπομονή, ανοχή και σεβασμό, διότι κατά κάποιο τρόπο καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει ε, την εξουσιοδότηση να διδάσκει τις άλλες χώρες. Υπάρχει όμως και το άλλο επίπεδο, το ελάχιστο κατόφλι σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία υποδεικνύονται από την ε, Διεθνή Δήλωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και κάτω από αυτό το κατόφλι κατά εμέ είναι αδύνατο να πάει κανείς. Και γύρω από αυτό το κατόφλι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πολύ ισχυρή και πολύ απαιτητική εποπτεία. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς καταφέρνουμε εμείς την πράξη να ασκήσουμε αυτούς τους ευφύης όρους. Τι πρακτικές μπορούν να μας υποδείξουν. Στην ε, πείρα που έχουμε από πλευράς Ιταλίας, εμείς προσπαθούμε να εισαγάγουμε ένα κριτήριο μέσω του οποίου όταν θα πρέπει να κυρωθούν διμερείς συμφωνίες μεταξύ της χώρας μας και χωρών που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακολουθούμε μια νέα πρακτική σε πειραματικό στάδιο να δεσμεύεται η κυβέρνησή μας τη στιγμή της κύρωσης της συμφωνίας να ξεκινά τις διαδικασίες καταγγελίας της ε, σύμβασης εάν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη χώρα εταίρων. Έχουν ξεκινήσει τρεις τέτοιες διαδικασίες. Μία συμφωνία με την Κίνα καταρχάς ε, για την κινηματογραφική βιομηχανία, δηλαδή σε πολιτιστικό επίπεδο. Μία συμφωνία η οποία έμεινε στάσιμη για πάρα πολύ καιρό στο Κοινοβούλιο, διότι υπήρχε μια σοβαρή ένσταση για το κατά πόσον μπορούμε να εμπιστευτούμε την Κίνα σε θέματα ε, λογοκρισία στον κινηματογραφικό τομέα και αποφασίσαμε να συνεχίσει η διαδικασία μέσω αυτής της ρήτρα και μια αντίστοιχη ρήτρα εφαρμόστηκε σε δύο πρόσφατες συμφωνίες τις οποίες κυρώσαμε, μία συμφωνία με το Μαρόκο για τη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο, πολύ ευαίσθητος ε, τομέας ε, μάλιστα σε, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην ε, Αφρικανική Ήπειρο και επειδή ακριβώς υπάρχει και ανοιχτό το θέμα των Σαχραουή και της Δυτικής Σαχάρας και το ίδιο φυσικά κάναμε και στη συμφωνία με το Κατάρ για αντίστοιχους λόγους. Θεωρώ λοιπόν ότι Ίσως η συγκεκριμένη ρήτρα, ε, θα δούμε κατά πόσον θα αποδειχθεί αποτελεσματική, αποτελεί έναν ενδιαφέροντα τρόπο ώστε να κατανοήσουν οι φίλες κυβερνήσεις με τις οποίες θέλουμε να έχουμε εταιρική σχέση, ότι ναι μεν τίνουμε χείρα βοηθείας, αλλά είναι και απαιτητική αυτή η χείρα, διότι απαιτούμε ένα ελάχιστο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον σε αυτό το απαραίτητο κατόφλι. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ. Όχι, ο κύριος Ταβάρης. Ε, Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα πρέπει σε λίγο να πάω στην συνεδρίαση της Επιτροπής μου για ψηφοφορία. Θα ήθελα ωστόσο να πάρω το λόγο και σημείωσα όλα όσα είπε ο Επιτροπός και ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Το βασικό θέμα, η λέξη κλειδί, είναι η ρεσιμότητα. Μιλάμε για κυρώσει σε περίπτωση που κρυθεί απαραίτητο, σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. αυτή η ευφυής ε, ερεσιμότητα ίσως να είναι καλύτερα από ότι η τυφλή ερεσιμότητα. Άρα μάλλον μου αρέσει αυτός ο νέος όρος. Ωστόσο θεωρώ ότι συχνά παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. Συχνά ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να τελειογήσει τα πάντα και οι βουλευτές εδώ μας ανέφεραν ότι δεν δίδεται ανθρωπιστική βοήθεια σε δικατορίες, για, για παράδειγμα. Αλλά ακούμε και το αντίθετο, ότι δεν διακινδυνεύεται σε καμία περίπτωση η ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια, δεν υπάρχει επαρκής ανεκτός χαρακτήρας, αν θέλετε. Μας είπατε ότι υπάρχουν νέοι και όλα αυτά θα πρέπει να λεφτούν υπόψη. Νομίζω όμως ότι Ακριβώς αυτό λείπει. Εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διερχόμαστε μία περίοδο κρίσης που μας αποδυναμώνει και αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει για την τήρηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Εκ παραλλήλου, θα πρέπει να είμαστε σημαντικά πιο συγκεκριμένοι από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωση για το τι θα πρέπει να τίθεται ως προϋπόθεση. Άρα, δεν μπορούμε να κρύβουμε τίποτα από τον φορολογούμενό μας. Η κρίση δεν έχει καταφτάσει ακόμα σε ό,τι αφορά θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο κόσμο. Κλείνοντας, τρία σχόλια θα ήθελα να κάνω. Με τους νέους αυτούς ε, όρους κλειδί που αναφέρατε, Ίσως να χάνονται οι στόχοι της πολιτικής μας. Η συνάδελφος Μπάιρ το είπε. Η πολιτική αλληλείας συχνά πατυχαίνει το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει με την αιρεσιμότητα. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τη γεωργία. Όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, στην Αραβική Άνοιξη δεν κάναμε απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Είχαμε πρόσφυγες από τα Βαλκάνια ή από την Ουγγαρία. Το 56. Εδώ όμως η Ευρώπη έλαμψε για τις απουσίες της. Και θα ήθελα οι εθνικοί βουλευτές να ξέρουν ότι είχε ψηφιστεί πρόγραμμα για τους πρόσφυγες, αλλά δεν είχε δώσει ως τώρα το πράσινο φως στο Συμβούλιο. Άρα λοιπόν κάτι θα πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική για τους πρόσφυγες, σε ό,τι αφορά τους εταίρους μας από την άλλη πλευρά της Μεσογείου. Να δούμε όμως τι κάνουμε και εδώ. Μέσω του Κοινοβουλίου θα πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρχει εφαρμογή και εποπτεία της εφαρμογής των όσων αποφασίζονται στα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμέλησε το καθήκον αυτό. 6 εκατομμύρια ευρώ αφορά το ζήτημα αυτό. Αλλά ανακύπτει και θέμα ηθικής ε, τάξης. Πώς μπορούμε να θεωρούμε ότι αποτελούμε φορέα ηθικής τάξης όταν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τις ίδιες αξίες. Ύστερα μιλάμε για θέματα μη ανάμειξης. Όλα αυτά συμπεριλήφθηκαν στο χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμω το αντιμετωπίζουμε κατά διαφορετικό τέλος. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία πιο συνολική προσέγγιση και πιο επικριτική αν θέλετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξαγάγουμε συμπαράσματα, όχι όπως είπε ο Ιταλός συνάδελφος, για παράδειγμα στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία, γιατί από εκεί μπορούμε να μάθουμε πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ τώρα. Να σας ε, σημειώσω ότι άλλοι έξι ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι λοιπόν. Um, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια αυτό που είχαμε κατά το παρελθόν, τη στενή συνεργασία με το καθεστώς της Λιβύης, Λιβύης ε, και το γεγονός ότι ε, χορηγήθηκαν χρήματα σε εξαγωγής όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο. Νομίζω ότι όπω ακριβώς και η ρεσιμότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το θέμα είναι πώ προχωράμε. Το κάνουμε με τη μορφή του εκβιασμού ή με τη μορφή διαλόγου, πολιτικού διαλόγου, όπου βεβαίω ε, και ερχόμαστε σε επαφή με τι κοινωνίε ε, των πολιτών και με τα κράτη-μέλη. Εκείνο που πρέπει να είναι σαφέ είναι ότι δεν πρέπει να βλάψουμε του πιο φτωχού με την αιρεσιμότητα. Γιατί πολλές φορές εμφανίζεται η κυβέρνηση η οποία περικόπτει την ελευθερωτική και μετά εμεί δεν δίνουμε χρήματα και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε χρήματα στην κυβέρνηση, δεν δίνουμε χρήματα και στους φτωχούς. Ε, ίσως πρέπει κανείς να σκεφτεί και τα κανάλια της διόδους. Πάντως, Συμφωνώ με αυτά που είπαν και άλλοι ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Αξιόπιστοι στη στρατηγική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν ε, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο παράδειγμα. Ε, μιλάμε για την Συμφωνία Αλίας με το Μαρόκο, παραδείγματο χάρη, όπου δεν ζητήσαμε καν ε, νομική γνωμοδότηση για το θέμα αυτό αναφέρθηκε ο συντονισμός και η συνέπεια στην πολιτική μας, όπως είπε και ο επίτροπο, ε, Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει καλύτερα να δούμε και την αιρεσιμότητα σε σχέση με εμάς, όχι μόνο για τους άλλους. Ε, επιβάλλουμε την αιρεσιμότητα σε χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά να δούμε και τι προσφέρουμε σε εμά. Παραδείγματο χάρη, ε, η βοήθεια που χορηγούμε ή να είμαστε συνεπείς για την ανάπτυξη, ε, να στηρίζουμε τη γεωργία, ε, τον κοινωνικό τομέα, να ωφελούνται οι πιο φτωχοί, να δεσμευτούμε για την κλιματική αλλαγή που περιπλέκει πολλά προβλήματα και θα πρέπει να είναι και η ερεσιμότητα για μας ε, με την έννοια ότι να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και στα χρήματα, τα κονδύλια που χορηγούμε αλλά και στον τρόπο που λειτουργούμε. Αναφέρθηκε και το θέμα των εμπορικών συμφωνιών. Εμείς μόνοι μας βάζουμε εκεί θέματα που οδηγούν σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι απαράδεικτο. Ε, θα πρέπει ε, να έχουμε ε, δίκες εμπορικές συμφωνίες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε εμπορικές ανταλλαγές ή αν θέλετε συμφωνήσει οικονομικής ε, συνεργασίας. Ε, και αυτό με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποκτήσουμε καλύτερη πρόσβαση ε, στους πόρους και εδώ θα ήθελα να φερθώ και σε αυτό που είπε η συνάλφος από την Αυστρία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Φέζο. Obrigada. Ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση ως τώρα. Και ήθελα να επανέλθω σε ένα από αυτά τα θέματα σχετικά με το τι γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Πορτογαλία εξετάζει το θέμα της ρεσιμότητας και φαίνεται ότι πάντα γίνεται αντιληπτή με αρνητικό τρόπο η ερωσιμότητα. Είναι δύσκολο να προσπαθήσουμε να δώσουμε την, ε, τον όρο, τον αρνητικό όρο της αιρεσιμότητας και αυτό νομίζω δυσκολεύει την εφαρμογή της αιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά και ένα πολυμερές επίπεδο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει διδάγματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία πριν από ένα-δύο χρόνια ψήφισε μία στρατηγική με το όνομα Ασφάλεια και Ανάπτυξη. Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουμε να διαβιβάσουμε. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια ούτε αντίστροφα. Εργαζόμαστε λοιπόν σε στρατηγικούς τομείς, συνεργαζόμαστε σε στρατηγικούς τομείς και προσπαθούμε να καταστρώσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τέσσερα υπουργεία. Φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν το α και το ω η προώθηση του κράτους δικαίου, οι στόχοι της χιλιετίας. Πρόκειται για αρχές τα οποία, οι οποίες διέπουν και δίνουν δομή σε όλες μας τις εργασίες. Τώρα, στο θέμα του τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην συζήτηση αυτή τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί μιλάμε για συνεργασία, για εξωτερική πολιτική και όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια των κυβερνήσεων. Οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που έχουν θεσμικές αρμοδιότητες στον τομέα αυτό. Άρα ερωτώ πώς μπορούν να μεταφερθούν κάποιες από τις αρμοδιότητες αυτές στα εθνικά κοινοβούλια. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω από πλευρά Γερμανία τι γίνεται εκεί και να σας πω ότι στην παρούσα φάση στην αναπτυξιακή εργασία θέτουμε νέους ε, στόχους και μια νέα συγκέντρωση ε, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική. Ή πολύ απλά λέμε πώς μπορούμε ένα και ένα να μην ε, ισούνται με δύο αλλά με τρία πώς μπορούμε να βρούμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Και άρα επικεντρωνόμαστε στον τομέα των ε, χωρών εταίρων, όχι μόνο σε 120 122 χώρες, αλλά σε 50 χώρες. Και παράλληλα, με το 0,7% του ΑΕΠ θέλουμε να πετύχουμε διπλασιασμό της αναπτυξιακής βοήθειας, άρα τετραπλασιασμό για τις 50 αυτές χώρες της αναπτυξιακής βοήθειας. Με άλλα λόγια, έχουμε πολύ καλύτερη και πολύ αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις χώρες αυτές, γιατί μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν πολύ πιο πολλά. Αυτό συνδέεται και με κάποιους όρους. Την άνοιξη αυτή ψηφίσαμε ένα νέο έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην γερμανική ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια της ε, Γερμανίας, όπου αποτυπώνται τα βασικά μας, οι βασικές μας αρχές. Και για παράδειγμα, εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι ως προς την αρνητική ρεσιμότητα, με κάποιες χώρες ε, όπου δεν είναι καλό το επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν ε, συνεργαζόμαστε σε ορισμένα επίπεδα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τον προϋπολογισμό για την άμεση βοήθεια και χρηματοδότηση κάποιων θεσμικών οργάνων εκεί. Για παράδειγμα, επίσης, ε, προσπαθούμε να αποτρέψουμε ε, περαιτέρω επιδείνωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εδώ ακούσαμε το θέμα της Ουγκάντα, της αντικής καταδίκης των σεξουαλικών μειονοτήτων ή έξι χρόνια φυλάκιση για κάποιον που είναι ομοφιλόφιλος από πλευράς μας. Όλα αυτά δεν ε, μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Δηλώσαμε λοιπόν στην Ουγκάντα ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος θα σταματήσουμε την δημοσιονομική βοήθεια Και όταν επιμείναμε, τελικά αποσύρθηκε η πρόταση νόμου. Ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Τώρα, για τα κίνητρα προσπαθήσαμε στη Βοζαμβίκη, για παράδειγμα, τα ελλείμματα τα οποία υπάρχουν στον τοπικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την δημοκρατική βασική οργάνωση, για παράδειγμα στην Ήπεθρο, να τα αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα λοιπόν αυτά. Θελήσαμε να δρομολογηθούν αυτό δεν ελήφθη επαρκώς υπόψη. Όταν όμως ε, ήρθε η απειλή της διαγραφής βοήθειας στον προϋπολογισμό, ήταν, ήταν έντονη η ανταπόκριση και τελικά συμφωνήσαμε. Άρα, αν υπάρχει θέληση, υπάρχει και αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό οι δωρητές ενός κράτους τα διάφορα υπουργεία. Είτε είναι υπουργεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε είναι υπουργεία ανάπτυξης, θα πρέπει να συντονίζουν τη δράση τους στην εκάστοτε χώρα. Αλλά υπάρχει ανάγκη και καλύτερου συντονισμού στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχουμε το καλό παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 απείλησαν την Κένια με οικονομικές κυρώσεις και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε αναπτυξιακή βοήθεια μεγάλου ύψους. Αυτά δεν μπορούμε να ε, επιτρέψουμε να συνεχιστούν. Ε, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλοι φορείς και ένα θέμα που συγκαταλέγεται σε αυτά είναι και το πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέματα διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο για μας η διαφθορά. Δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα κατά της διαφθοράς, αλλά θα μπορούσαμε να θέσουμε μια απέτηση ως προς την διαφθορά, γιατί τελικά αν τα κονδύλια αναπτυξιακής βοήθειας καταλήγουν στα χέρια διαφθαρμένων κυβερνήσεων, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε την βοήθεια αυτή έναντι του φορολογούμενου. Οι διεθνώς ε, δραστηριοποιούμενες ε, εταιρείε και αυτές θα πρέπει πολύ πιο έντονα να ζητούν και να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις θηγατρικές τους ε, εταιρείες στις ξένες χώρες. Γιατί και εδώ σημαίνει πολλά και μπορεί να εφαρμοστεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λοκπίλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στα θέματα τα οποία έθιξε η κυρία Μπάιερ, τα οποία τα συζήτησε και προηγουμένως και επαναλήφθηκαν και από άλλους συναδέλφους μας. Είπατε ότι υπάρχει ένας κοινός ορισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το ζήγισμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αυτό όχι μόνο με τους εταίρους μας, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι αυτό δεν αποτελεί καλή κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να υπάρχει προτεραιότητα ότι τα πρώτα δικαιώματα είναι τα αστικά, τα προσωπικά, τα ατομικά δικαιώματα και μετά έρχονται τα κοινωνικά και τα εργασιακά. Νομίζω ότι μας έχει σημαντεύσει στην Ευρώπη ο ψυχρός πόλεμος, αυτή η ιδεολογία. Και αν αποτυπώνεται αυτό στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι σαφές ότι και οι δύο κατηγορίες προαπαιτούν η μία την άλλη. Μόνο έτσι μπορεί ο κόσμος να είναι ελεύθερος και να μην φοβάται και έτσι να ζει. Αυτές είναι οι δύο κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι βασικό λάθος αν θέτουμε μια τέτοια ιεράρχηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο η τρίτη γενιά, το δικαίωμα ανάπτυξης, ομολογώ ότι δεν έχει ε, επεξηγηθεί τόσο καλά όσο οι άλλες γενιές. Δεν έχω πολλά άλλα να προσθέσω σε αυτά που ακούσαμε σε ό,τι αφορά τους όρους που θα πρέπει να θέτουμε αν ε, υπάρχουν τόσο μεγάλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα για τις σεξουαλικές μειονότητες θα πρέπει στους τομείς αυτούς να συνεργαστούμε ακόμα πιο πολύ με τους μη κρατικούς φορείς και δεν εννοώ μόνο τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εννοώ για παράδειγμα μεγάλες θρησκευτικέ οργανώσεις οι οποίες κατά κανόνα και αυτές με πολύ περιορισμένο τρόπο κατανοούν την ανθρώπινη ταυτότητα και δεν συμπεριλαμβάνουν θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε επιρροή και στις μεγάλες αυτές οργανώσεις ακόμα πιο πολύ ως τώρα. Αυτό ως απάντηση στην κυρία Μπάιερ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Γκόμες. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε όσοι εργαζόμαστε στον τομέα τη ανάπτυξη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρί καλή κυβέρνηση, χωρί κράτος δικαίου, χωρί ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά πρέπει να συνάδουν. Και περιλαμβάνουν και τα θέματα διαφθορά, γιατί η καλή κυβέρνηση συνεπάγεται την καταπολέμηση τη διαφθοράς. Το πρόβλημα είναι ότι όλε αυτέ οι έννοιε έχουν ε, καταλήξει, αν θέλετε, στο περιθώριο προ όφελο λέξεων και έννοιων που δεν περιλαμβάνουν την καλή διακυβέρνηση, δεν περιλαμβάνουν την ομαλή μετάβαση στην δημοκρατία. Πολλές κυβερνήσεις που βρίσκονται σε φάση μεταβατική και οδεύουν προς την δημοκρατία απλά θέλουν την νομιμοποίηση, την νομιμότητα για την ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες οργανώσεις. Μου αρέσει ο όρος και η έννοια της έξυπνης, της ευφυούς ρεσιμότητας. Στην αλήθεια όμως ούτε ευφυής είναι, ούτε ρεσιμότητα είναι. Δεν προωθεί κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Αντιθέτως, ένα σχέδιο δημοσιονομικής αρρωγής κατά το παρελθόν. Τι συνέπεια είχε μια τυφλή ρεσιμότητα. ή μη ερεσιμότητα σχεδόν και ουσιαστικά τα κριτήρια όπως ε, υπέδειξαν κάποιοι συνάδελφοι είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, πολύ βασικά. Όταν μιλάει κανείς για παράδειγμα κατά της κυβέρνησης και φυλακίζεται, πρόκειται για παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων. Αν μου πάρουν τη γη μου για να χτίσουν το οτιδήποτε για τον ε, οποιοδήποτε ε, πολιτικό πρόκειται για παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων. Είναι καταφανή αυτά τα περιστατικά. Κάποιοι συνάδελφοι ρώτησαν τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Θέλω να πω ότι η αρχή της ρεσιμότητας υπάρχει ως μέσο και είχαμε αναρωτηθεί αν θα πρέπει να περιοριστούμε και να επικεντρωθούμε στην δημοσιονομική βοήθεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε ακουστεί ως επιχείρημα ήταν σε ανταγωνιστική φάση με την Κίνα σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Όμως τι κρυβόταν πίσω από αυτή την ανταγωνιστικότητα. Γίνεται μια απόπειρα νέων αποκαικρατικών δεσμών για να αποδώσουμε κέρδους, κέρδους για λίγα άτομα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι η Κίνα βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και θα πρέπει να έχουμε θα πρέπει να διδαχτούμε από τα παθήματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να διδαχτούμε από την Αραβική Άνοιξη. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε ό,τι αφορά τις επαφές μας με τις άλλες κυβερνήσεις. Θα πρέπει να διοχετεύουμε τα κονδύλια στην κοινωνία που τα χρειάζεται. Και υπάρχουν άλλες χώρες και υπάρχουν κοινωνίες, κοινότητες που περιμένουν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα, τα οποία όμως εμείς τα δίνουμε ως δημοσιονομική βοήθεια στις κυβερνήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την Ερυθρέα. Θα πρέπει να γίνει έρευνα επιτόπου και είναι σοβαρή η περίπτωση αυτή γιατί εμπλέκει και έναν πολίτη σουητικής υπηκότητας. Ας δούμε τι γίνεται σε άλλα κοινοβούλια, σε αφρικά, αφρικανικά κοινοβούλια. Ας δούμε τι γίνεται για την με την Αιθιοπία. Η Αιθιοπία, ξέρετε, δεν είναι μια τυχαία χώρα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Αφρική. Είναι η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ότι δεν βλέπει τις τεράστιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ας δούμε τι έγινε το 2005, τι έγινε το 2010. Η κατάσταση πραγματικά προκαλεί φρίκη. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά και την επίλυση συγκρούσεων. Και αυτό αναφέρθηκε. Τα προβλήματα της ε, Αιθιοπίας και της Ερυθρέας συχνά αφορούν αναπήλυτα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα σύνορα. Μία ερώτηση. Ας δούμε για παράδειγμα την περίπτωση της Αγγόλας. Ναι, η πρόεδρος λέει παρακαλώ να, να σεβαστείτε το χρόνο που έχει στη διάθεσή σας. Τι έγινε με τους νεαρούς φυλακισμένους στην Αγγόλα. Τι κάναμε να εξετάσουμε το θέμα τους. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο ομιλίας, διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο άλλοι συνάδελφοι. Ο κύριος Νεοφίτου τώρα και στη συνέχεια ο κύριος Κάσμαρη και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα. Και σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε για τη διοργάνωση αυτής της συνάντησης για το σημαντικό θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας συμφωνούμε απόλυτα πάνω στην βασική αρχή ότι είναι αδιανόητο σε μια χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα την ίδια στιγμή να δίδεται αναπτυξιακή βοήθεια σε ένα διεφθαρμένο και δικτατορικό καθεστώς που στο τέλος αυτά τα λεφτά αντί να πηγαίνουν για την αναπτυξιακή πολιτική ε, χρησιμοποιούνται για προσωπική χρήση από τους δικτάτορες. Όμως την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι όσο πιο δικτατορικό είναι ένα καθεστώς, τόσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα φτώχειας στην χώρα. Και αυτοί οι αδίστακτοι δικτάτορες δεν γνιάζονται για την φτώχεια των πολιτών. Εξού και δεν γνιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Άρα ακολουθώντας την σωστή αρχή ότι δεν δίνουμε αναπτυξιακή βοήθεια εκεί που υπάρχουν δικτατορικά καθεστώτα, στο τέλος αυτοί που πληρώνουν το κόστος αυτής της σωστής πολιτικής ε, είναι οι απλοί πολίτες. Μήπως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και την περίπτωση που θα μπορούσαν να δοθούν σημαντικά κίνητρα σε ευρωπαϊκές εταιρείες για δραστηριοποίηση σε αυτές τις χώρες, για αναπτυξιακούς σκοπούς, για να επενδύσουν και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίες και θα βοηθήσουν και την κοινωνία αλλά και τους πολίτες αυτών των χωρών. Κάτι παρόμοιο γνωρίζουμε ότι εφαρμόζεται και από την Κίνα και έχει και τα θετικά της αποτελέσματα και για την οικονομία της Κίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κάσμαρεκ, ο οποίος θα μας διαβάσει μια επιστολή εκ του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ κύριε Κάσμαρεκ, έχετε το λόγο και κατόπιν θα δώσω την, κυρία, την προεδρία στην κυρία Λοκπίνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε στην Πολωνία είχαμε προεδρικές ε, κοινοβουλευτικές εκλογές, γι' αυτό και δεν μπορούν να παραστούν οι Πολωνοί βουλευτές. Έχω όμως ε, μία επιστολή του Προέδρου ε, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πολωνικού Κοινοβουλίου, την οποία και σας διαβάζω. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς και την Επιτροπή σας για την πρόσκληση ε, για την ε, συμμετοχή στη διακυβερνητική συνεδρίαση της 11ης Οκτωβρίου. Δυστυχώς, λόγω των προεδρικών ε, και βουλευτικών εκλογών στην Πολωνία, δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω. αλλά ως εκπρόσωπος του Πολωνικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σε εκφράσω την πεποίθησή μου ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και καθόλου επίκαιρο. Το θέμα της αιρεσιμότητας είναι ένα σημείο που αφορά και την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Έγινε και μια σχετική σύνοδος επί του θέματος στη Βαρσοβία. Οι Πολωνοί βουλευτές ε, κάνουν το καθήκον τους και προσπαθούν να προωθήσουν ε, τα δημοκρατικά δικαιώματα προς Ανατολή, Λάς, ιδίως στη Λευκορωσία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τα προγράμματα αυτά σε χώρες στις οποίες παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο μέλλον θα μπορέσουν να δημιουργήσουν και να βοηθήσουν στη δημιουργία δημοκρατικών θεσμών στις χώρες αυτές πέραν των σωνόρων της χώρας μου, πάντα είμαι υπέρ των ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, ζητούν να υπάρχει αυτή υπό όρους ε, ε, εκχώρηση δικαιωμάτων. Ήμουνα παρόν σε μια απεργία στην οποία συναντήθηκα με τους εκπροσώπους ε, ε, της απεργίας αυτής στο Καζακστάν. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια καταδίκη για τα όσα γίνονται από πλευράς κυβέρνησης όταν ε, κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε θεωρώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα χρειαζόμαστε μια δημοκρατική κοινωνία και αλληλεγγύη στην κοινωνία αυτή. Υπάρχει ακόμα λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας. Η Κίνα επί παραδείγματι είναι οικονομικός εταίρος αλλά δεν είναι εταίρος μας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο όσον αφορά και τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αλλά δεν σκέφτεται κανείς να σταματήσει τις οικονομικές σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες. Όσον αφορά τώρα την Κροατία, η οποία ολοκληρώνει τη διαδικασία προσχώρησή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκα με Σέρβους και Κροάτες εκπροσώπους και μιλήσαμε για τις ε, σειράξεις και τις συγκρούσεις που είχαν στο παρελθόν οι λαοί αυτοί. Αλλά θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη και τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες αυτές. Πώς μπορούμε να μιλάμε για παραβίαση των δικαιωμάτων ε, χωρίς να φοβούμαστε ότι μπορεί να διακυβεύονται και οι οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις στις χώρες στις οποίες πλήχθηκαν ε, από διάφορα προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό καθήκον, ένα καθήκον για την εξωτερική υπηρεσία ε, ε, εξωτερικής δράσης και θα πρέπει να μιλάμε με πιο δυνατή και πιο σαφή φωνή για το τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις. Η αιρεσιμότητα μπορεί να είναι δύσκολη στην πράξη, αλλά σε θέματα συνεργασίας, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ε, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όταν η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σοβαρή, δεν μπορούμε ε, να πούμε ότι δεν θα δίνουμε την κατεπίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Θα πρέπει να δίνονται κυρώσεις ανάλογα με τα ε, προβλήματα που υπάρχουν και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να εξετάσουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ελπίζω να μπορέσουν να τα Σας εύχομαι καλή δουλειά σε αυτή την κοινοβουλευτική συνεδρίαση που θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ε, ε, συνεργασία μεταξύ εθνικών ε, κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μπορέσω να σας συναντήσω σύντομα στις Βρυξέλλες ή στη Βαρσοβία. Ο Ρέσατ Κάλλη ε, έστειλε αυτή την επιστολή, εκπρόσωπο τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ρέσατ Κάλλη σαφώ ε, θα παραστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και ξαναδίνω το λόγο στους ε, Πολωνούς ε, συναντελφούς ε, να τους πω ότι βεβαίως και αν έχετε εκλογές δεν μπορείτε να είσαστε εδώ. Αναλαμβάνω τώρα εγώ πλέον την Προεδρία εδώ στη συνάντησή μας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους από τα Εθνικά Κοινοβουλία εξ ονόματος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη συνάντηση με την Επιτροπή Ανάπτυξης μετά τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Ως ε, πρώτο θέμα έχουμε τη σχέση ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Παλαιότερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχαμε δύο φορές συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια. Ε, τη μία φορά οι συναντήσει αυτέ έλαβαν χώρα στο Βερολίνο και την άλλη στις Βρυξέλλες και ω Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπιστώσαμε ότι δεν είναι εύκολο να έχει κανείς την σωστή οργανωτική δομή γιατί στα διάφορα κράτη ε, υπάρχουν και διαφορετικές ε, προσεγγίσεις. Η πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντάσσεται σε διάφορες άλλες πολιτικές, μερικές φορές και στην πολιτική της μετανάστευση. Στον πρώτο γύρο ακούσαμε το κατά πόσον ε, η αιρεσιμότητα, όπως λέγεται, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να έχει ε, να επιδράσει την ε, αντιμετώπιση της ένδυας. Εγώ δεν άκουσα κανένα επιχείρημα ε, προς την κατεύθυνση του ότι υπάρχει αντίφαση. Αυτά, αυτό ήθελα απλά να πω συμπερασματικά. Τώρα λοιπόν στο δεύτερο γύρο έχουμε το θέμα του κατά πόσον η αιρεσιμότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ένα περιβάλλον πολλών δωρητών. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να θίξουμε το εξή θέμα. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της αιρεσιμότητας τι εργαλεία έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να έχουμε ε, πολιτικές ε, που να προσανατολίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα βρούμε και τις απαντήσεις. Ακούσαμε προηγουμένως, αλλά θα επανέλθουμε, ότι υπάρχει ένα ειδικό μέσα στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, αυτή η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις συμφωνίες αναπτυξιακής βοήθειας με τις τρίτες χώρες. Εναπόκειτο λοιπόν σε εμά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουμε έλεγχο για το κατά πόσο αυτές οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφαρμόζονται ή όχι. Ε, και τώρα ε, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ε, συμφωνίες που συζητούνται, η εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο και η άλλη με την Κολομβία. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να ακούσω από εσάς ε, το πώς ακριβώς η αιρεσιμότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, προβάλλεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, ε, στη συζήτηση θα πρέπει να εξετάσουμε και τα διάφορα επιχείρηματα κατά της αιρεσιμότητας, όπως ασύμμετρες σχέσεις ανάμεσα στους δωρητές και τους δικαιούχους, αυθαίρετες αποφάσεις, πολιτικά και άλλα συμφέροντα που υπάρχουν. Ε, ιονή ε, αναποτελεσματικότητα και τέλος ε, ε, διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Όπως και στον προηγούμενο γύρο συζητήσεων, παρεμβάσεων, θα έχουμε ίσως ένα ή δύο μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Τσίμα, η οποία ζήτησε τον λόγο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την παρέμβασή της. Η κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα αυτά τα θέματα που ετέθησαν λιγάκι όπως έκανα και κατά τον πρώτο γύρο να τα συμπληρώσω και τώρα με έτσι μια, ένα προκλητικό αίτημα. Δηλαδή το θέμα της ερεσιμότητας των ε, συνθήκων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να το δει κανεί και από την άλλη πλευρά του νομίσματο. Όχι δηλαδή πώ ακριβώ εφαρμόζονται τα κράτη-μέλη στι χώρε εταίρου, αλλά να τεθεί και το ερώτημα πώ ακριβώ συμβάλλουμε εμεί με τι ε, συνθήκε μα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από εμά ε, από τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να παραπέμψω στο ότι παραδείγματο χάρη ο Λιβιέντε Σούτα, ο ειδικό απεσταλμένος για θέματα επισητιστική ασφάλειας, απέτυχε στην προσπάθειά του να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν έτσι ώστε όλες οι εμπορικές συμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνάπτονται με αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν μια ρήτρα όπου θα απαιτείται οι συνθήκες να ελέγχονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους για το δικαίωμα στην διατροφή, σε τρόφιμα. Αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν λέει ότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει και δεν το επιθυμούμε. Ε, δεν είναι δηλαδή δυνατόν να βλέπουμε ε, μέχρι ε, ποιου βαθμού παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμάς, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, οι συμβάσεις που συνάπτουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη, οι συμβάσεις αυτές να μην συμβάλλουν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και κυρίως ε, στις εμπορικές συμφωνίες πολύ συχνά έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κάτι άλλο που θέλω να θίξω επίσης ε, για να είμαστε έτσι και συγκεκριμένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσε μία πρόταση με βάση την οποία όλα τα κράτη ε, τα οποία δεν έχουν υπογράψει εμπορικές συμφωνίες ή δεν έχουν ε, αναστείλει τις συμφωνίες αυτές δεν έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τελική ανάλυση σε αυτά τα κράτη θα πρέπει να τους αρνηθούμε την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα κράτη αυτά οφείλουν ε, να φτιάξουν τη δική τους αγορά, να εμπορεύονται τα δικά τους προϊόντα και στη τελική ανάλυση, ανάλυση να ε, φροντίζουν ε, για την ψηφιστική ασφάλεια. Αν δεν το πράττουν αυτό, ε, πρόκειται για ε, παραβίαση της, του άρθρου 8 της Συνθήκης Λισαβόνας. Υπάρχει λοιπόν η παράκλησή μου και από την άλλη πλευρά των κρατών που και αυτά καλούνται να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν βλέπω κανείς άλλος να έχει ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να ξέρετε ότι έχουμε χρόνο για συζήτηση Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε ε, τα θέματα σε βάθος ε, και κατά τον πρώτο γύρο και τώρα άκουσα από την κυρία Τσίμα ορισμένες ερωτήσεις ε, και θα ήθελα να τοποθετηθείτε στο ποια ακριβώς είναι η θέση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Εδώ στο βήμα δεν έχουμε κανέναν άλλο για να μιλήσει επί του θέματος. Νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιον ο κύριος Βιλ Ντεβίλ από την ΔΕΦΚΟ. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να σας συστηθώ πριν κάνω μια απόπειρα να απαντήσω. Λέγομαι Jean-Louis Ville, είμαι ο Διευθυντής του Τμήματος ε, Διακυβέρνηση, Δημοκρατία και Κατεπήγοντα Θέματα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενική Διεύθυνση ε, για τη Συνεργασία. Μία πρώτη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, όχι για τη συζήτηση η οποία ανεξελίξει αυτή τη στιγμή, αλλά για τις παρεμβάσεις που μόλις ακούσαμε. Να σας πω ότι ως ε, ε, επικεφαλής ε, του τμήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμφωνώ απολύτως με τα όσα ακούσαμε. Δεν ε, εναπόκειται άλλωστε σε μένα να αμφισβητήσω κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ. Να επανέλθουμε τώρα στην ουσία, στο θέμα της αιρεσιμότητας. Νομίζω ότι πρόκειται για ανοιχτή συζήτηση. Η ποικιλομαρφία ε, των θεμάτων τα οποία ετέθησαν άλλωστε απαντούν από μόνα τους στο ίδιο θέμα. Το θέμα της ερετησιμότητας ε, δεν είναι τόσο το να γνωρίζουμε αν χρειάζεται ή όχι το να επιβάλλουμε έρους, αλλά το θέμα είναι με ποιον θα το επιβάλλουμε τους όρους, ε, θα τους επιβάλλουμε και πώς. Κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες ετέθησαν εδώ στην αίθουσα είναι ερωτήματα τα οποία θέτουμε και εμείς ε, οι ίδιοι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ε, εφαρμογή των ε, προγραμμάτων βοήθειας και συνεργασίας. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν από τους ομιλητές εδώ, νομίζω η Κάσμαρε και ο κύριος Στονίνη, αυτά επεσήμενα, είναι ότι χρειάζεται διάλογος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ε, επιδείξουμε φιδό στο διάλογο μεταξύ των ε, ε κυβερνήσεων των χωρών ε, που συμμετέχουν στη βοήθεια. Μπορεί βέβαια ο διάλογος όπως κάποιοι είπαν ε, ορισμένες φορές να είναι σκληρός και δύσκολος, μπορεί να είναι και διάλογος κοφών. Αλλά δεν έχει τόση σημασία. Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε την άποψή μας σε κάποιον τρίτο, ακόμα και αν έχουμε άποψη επί του θέματος. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο λοιπόν, ικανή και αναγκαία συνθήκη να γίνει ο διάλογος. Δεν μπορεί να περάσουμε στις κυρώσεις χωρίς προηγουμένως να έχουμε κάνει μια απόπειρα να ε, συνομιλήσουμε με τους εταίρους μας και να αντιπαρατεθούμε ακόμα. Ε, όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις ή μάλλον τα περιοριστικά μέτρα, θα τα αποκαλέσω έτσι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε γιατί είναι όλα ή τίποτα. Ή θα σταματήσουμε και επομένω εκεί πάβει η συνεργασία με την κυβέρνηση και τιμωρείται ο λαός. Ή αλλιώς δεν σταματάμε και θέτουμε τα ερωτήματα τα οποία εύλογα θέτεται αν θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Και εκεί νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω και ένα παράδειγμα για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή στη Ζιμπάμπιο, ε, όπως είπε ο Επίτροπος, βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ε, κυρώσεων ή περιοριστικών μέτρων αν θέλετε. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται τόσο και από πλευράς μας όσο και από πλευράς κυβέρνησης αλλά και κοινωνίας στη Ζιμπάμπουε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πλήρη αναθεώρηση της ε, κατάστασης Γίνεται βεβαίως με τις αρχές όπου διαφαίνεται κάποια συμφωνία για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, αλλά το κάνουμε και το κάνουμε ιδίως με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Διότι μέσω αυτής της οδού, κατά την άποψή μας, θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να οικοδομούμε τη μελλοντική συνεργασία και τη συνέχιση της συνεργασίας με τη χώρα αυτή. Αυτό που ισχύει για τη Ζιμπάμπουε φυσικά θα μπορούσε να ισχύσει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν θα ήθελα να κάνετε λάθος ε, και να φύγουν ε, οι βουλευτές που είναι παρόντες εδώ σήμερα με τη λανθασμένη άποψη ότι δίνεται μάχη μεταξύ διαφορετικών απόψεων, δηλαδή ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρεσβεύει τις ίδιες αρχές. Δεν θα πρέπει να χάσουμε το στόχο μας λοιπόν ε, και να έχετε λάθος στόχο. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή η οποία θα ε, υποβοηθήσει την έλλειψη μέτρων και κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δει πώς μπορούμε από κοινού να οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη καλύτερα την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων άκουσε επίσης κάποιες παρατηρήσεις για τις σχέσεις μεταξύ του τι δίνουμε εμεί προ τα έξω και τι θα έπρεπε να πετούμε ε, από τους υπολείπου. Αναφερθήκαμε στην ελευθερία του τύπου και σε μία σειρά άλλα παραδείγματα, τα οποία νομίζω ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτηση. Κατά την άποψή μου, ε, δεν έχει σημασία να πούμε ότι ας επιβραβώσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να δείξουμε και ποιες είναι οι δικές μας αδυναμίες για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να εκχωρήσουμε αρμοδιότητες και να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους συνομιλητές μας. Μια τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι όλα τα ζητήματα που ε, θίξατε σίγουρα αποτελούν αντικείμενο της αναθεώρησης ε, που η κυρία Άστον είπατε εκπρόσωπος ε, θα παρουσιάσει στο πλαίσιο τη εντολή τη, δηλαδή μια πλήρη αναθεώρηση τη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο μα έχουν υποσχεθεί και θα φτάσει. Δεν μπορώ σήμερα να σα πω ε, τι ακριβώς θα γίνει γιατί δεν είμαι εν γνώση του τι ακριβώς ετοιμάζει αλλά όταν θα φτάσει θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση. Ε, επίσης θα δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μελλοντικέ δημοσιονομικές ε, προοπτικές αλλά σίγουρα θα υπάρχει μια πτυχή που θα επικεντρωθεί στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και πέρα το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράσουν την απόψή τους για να πούν κατά πόσον θεωρείται επαρκή. Ε, η έμφαση που δίνεται ή αν χρειάζεται ε, τι περαιτέρω. Ε, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση η αν χρειαζεται τι περαιτερω αλλα αυτη ειναι μια συζητηση η οποια θα γίνει στο μέλλον. Αυτά μπορώ να σας πω από πλευρά ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς δεν έχω αρμοδιότητα για να σας απαντήσω εκ μέρου τη υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ich, äh, danke Ihnen für die Aus... Σας ευχαριστώ για τις ε, εξηγήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος αν μου επιτρέπετε, σωστά αναφέρετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε και περιμένουμε κατεπηγόντως σχέδιο αυτή της αναθεώρησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για όλα τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθεί μια επισκόπηση όλων αυτών των μέσων. Το περιμένουμε λοιπόν το έργο αυτό και καλωσορίζουμε το ότι η Λέδη Άστον δεσμεύτηκε να προβεί σε μια τέτοια εισβάθος επισκόπηση και φυσικά θα θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς ως Κοινοβούλιο στην συζήτηση αυτή. Για ένα θέμα θα ήθελα να σας απαντήσω. Δεν ξέρω μήπως ήταν θέμα γερμανικής ερμηνεία. Συζητήσαμε και πολλοί συνάδελφοι το έθεσαν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επικριτικοί για τις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς τις εφαρμόζουμε πίστη στις αρχές μας. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η αυτοομοιρία δεν ε, αποφέρει τίποτα. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπονόησαν οι συνάδελφοι. Όχι βέβαια, η αυτοκριτική όμως είναι κάτι το σημαντικό. Και θα ήθελα σε να επαναλάβω εκ νέου το εξή. Αν ασκούμε αυτοκριτική και κοιτάμε τα σφάλματα του παρελθόντος σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την τρομοκρατία, όπου, για παράδειγμα, υπήρξαν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι αυτό εννοούσαν οι συνάδελφοι, η κυρία Τεκάιζερ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ε, συμμετείχα στο πρώτο τμήμα της συζήτηση σήμερα το απόγευμα, οπότε υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά που θα πω να έχουν ήδη συζητηθεί. Αλλά ε, σας έχω εμπιστοσύνη, θα με προειδοποιήσετε εσείς σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να σταθώ σε μια φιλοσοφία η οποία ε, προκύπτει όλο ένα και περισσότερο στη συζήτηση που κάνουμε για τη αιρεσιμότητα, χρησιμοποιώντα σαν παράδειγμα τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ε, που συζητάτε με την Κολομβία και που αναφέρατε κι εσείς. Νομίζω ότι όλο και περισσότερο σε επίπεδο κοινοβουλίου και με τις νέες εξουσίες που δίνει η συνθήκη της Λισαβόνα σε θέματα διεθνούς ε, εμπορίου, έχουμε πλέον δικαίωμα συναπόφαση στο θέμα αυτό και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθεται ίσως λιγότερο για το κατά πόσο θα υπογράψουμε ή δεν θα υπογράψουμε γιατί η συγκεκριμένη χώρα έχει ε, αμφισβητήσιμα αποτελέσματα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο στο κατά πόσον μπορούμε εμείς μέσω συμφωνιών, επί παραδείγματι εμπορικών συμφωνιών, να οδηγήσουμε τη χώρα αυτή να κάνει τη βαθιά τομή που χρειάζεται. Δηλαδή, να γίνει μια αλλαγή στη χώρα και ενδεχομένως, εάν η χώρα αυτή αλλάξει, κατά πόσον μπορούμε, ε, εάν ε, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, να βάλουμε ένα φραγμό και να σταματήσουμε τη συμφωνία. Υπάρχουν δύο στιγμές λοιπόν, τη στιγμή της υπογραφής της συμφωνίας και από εκεί και πέρα την παρακολούθηση και την εφαρμογή κυρώσεων δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα εδώ, ε, αλλά είμαστε κάπου στη μέση. Και νομίζω ότι στη συμφωνία με την Κολομβία, η οποία είναι υποσυζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο άσχημα ε, περιστατικά υπάρχουν, δολοφόνιες, απαγωγές, ε, παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίες έχουν παρισφρήσει στο κυβερνητικό πλαίσιο. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Είναι ζωφερή η κατάσταση στην Κολομβία και είναι αλήθεια ότι εδώ και κάποια χρόνια και ιδίως ε, από τότε που ο πρόεδρος Ουρίμπε άλλαξε στάση, έχουν αλλάξει πράγματα και νομίζω ότι υπάρχει και η πίεση αυτής της συμφωνίας η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Και στην τελευταία αντιπροσωπεία ε, που έκανε το Κοινοβούλιο, στις τελευταίες αντιπροσωπείες, βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερους θυνικισμούς, ακόμα υπάρχουν βέβαια, υπάρχουν κάποιοι νόμοι για τις αποσημειώσεις των θυμάτων ε, και όταν ε, τα θύματα θεωρούνται ότι υπάρχουν ε, προβλήματα σε θέματα συλλογικά, ε, υπάρχουν κάποιοι νόμοι για την περιουσία, δηλαδή αλλάζουν κάποια πράγματα σε νομικό επίπεδο τουλάχιστον, τα οποία μένει να εφαρμοστούν. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε να δούμε κατά πόσον αυτά τα οποία ψηφίστηκαν και έχουν γραφτεί πλέον σε νόμο θα υλοποιηθούν και να φτάσει η στιγμή που να μπορέσουμε να πούμε ότι πλέον είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορούμε να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Κολομβία, αλλά πώς μπορούμε να επαγρυπνούμε και να γνωρίζουμε ότι θα τα τηρήσει όλα αυτά τα οποία ε, ανέλαβε να κάνει η Κολομβία ε, και τι μας προσφέρει η συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να επαγρυπνούμε. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται και το ερώτημα που θέτουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορούμε να πάμε στην Κολομβία και να τους πούμε ναι θα υπογράψουμε αλλά πρέπει να κάνετε το τάδε και το δίνα και να κάνετε και την επιπλέον πρόοδο. Θεωρώ ότι η Κολομβία είναι ένα καλό παράδειγμα. Ε, υπήρξε όλη αυτή η εξέλιξη και υπάρχει και εξέλιξη σε εμά ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές ομάδες, μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και θεωρούμε ότι έχουμε πλέον ε, μοχλούς ε, πίεσης για να αλλάξουν τα πράγματα και σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και αυτό βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο ε, πλέον ε, υπάρχουν υποσχέσεις και πλέον νομίζω ότι στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι συμφωνίες υπάρχουν κάποια όπλα που μας επιτρέπουν να ελέγξουμε τις συμφωνίες ώστε αυτή η αιρεσιμότητα να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι στο μέλλον ε, στο παρελθόν συγγνώμη, όπου παρέμεινε νεκρό γράμμα στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχω ε, στον κατάλογο των ομιλητών συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα θέλαμε να ανταλλάξουμε απόψει και με εσά από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Υπήρξε μια ερώτηση από την κυρία Ντεκάιζερ προς την ε, Επιτροπή ε, και θέλω να δώσω δυνατότητα στην Επιτροπή να απαντήσει, αλλά θέλω να σας ενθαρρύνω. Για μένα, παραδείγματο χάρη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω ε, κατά πόσον σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν συμφωνίες με την Κολομβία ε, και πώς ε, το αντιμετωπίζετε σε αυτό. Υπάρχει τώρα ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το κατά πόσον υπάρχει σύστημα ελέγχου στην περίπτωση ε, κατά την ε, οποία η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει συμπεριληφθεί στη συμφωνία με την Κολομβία. Παρακαλώ, έχετε και πάλι το λόγο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας ε, για την αναγνώριση των σφαλμάτων. Όταν υπάρχει διάλογος δεν μπορεί να συνεχιστεί αν δεν αναγνωρίζει ο ένας ότι άσφαλε ενώπιον του άλλου. Στην ερώτηση της κυρίας Ντεκέιζερ για το μοχλό Πολύ σωστά το περιέγραψε. Νομίζω σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια εμπορική συμφωνία, αλλά μπορούμε ε, να εφαρμόσουμε τον ίδιο μοχλό πίεση σε ένα μέσο διαρθρωτικής ε, υποστήριξης σε περίπτωση που υπάρχουν και κάποια θέματα κονδύλια στον προπολογισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαδικασία μπορεί να υπάρχει μία απεικόνηση της αρχικής κατάστασης που μας περιγράφει μία ζωφερή, πολύ ζωφερή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε και κατά πόσον τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλή πίωση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι το είπε και ο Επίτροπος. Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη ε, με την ε, τάδε τη δίνα χώρα. Δεν έχει σημασία τόσο η χώρα. Δεν έχει σημασία το να μπορούμε να πούμε ότι αν δεν κάνετε αυτό ή αν δεν κάνετε το άλλο η κατάσταση θα αλλάξει εκ βάθρων ε, και μάλιστα πολύ ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί σας αλλιώς θα σας επιβάλλουμε κυρώσεις. Δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση εν εξελίξη. Σας το είπα και προηγουμένως, ένα από τα μέσα τα οποία έχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Διότι θεωρούμε ότι μέσω εσωτερικής πίεσης προς τις ε, ε κυβερνήσεις θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δυστυχώ δεν γνωρίζω τα τη ε, συμφωνία με την ε, Κολομβία. Νομίζω ότι η κατάσταση που μα παρουσίασε η κυρία Ντεκέιζερ είναι πολύ πιο πλήρη από τι πληροφορίε που μπορεί να έχω εγώ. Αλλά το σκεπτικό είναι το εξή. Όταν υπάρχει ένα μηχανισμό εποπτεία, παρακολούθηση, συνέχεια ή όπω θέλετε αποκαλέστε το τη κατάσταση, ε, είναι κάτι το οποίο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την έννοια ότι κάθε αντιπροσωπεία κάνει μία ε, τακτή αναθεώρηση της κατάστασης σε ένα χώρα και από εκεί και πέρα λαμβάνει υπόψη ε, τις θετικές ή τις αρνητικές εξελίξεις σε κάθε χώρα. Τα μέτρα υποπτίας μπορεί να υπάρχουν, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι παραμέτρους θα λάβουμε υπόψη. ποιους τομείς πρέπει να εξετάσουμε, ποιες συμβάσεις πρέπει να κυρωθούν ή οτιδήποτε άλλο. Ε, άλλο το μέτρα, άλλο η σύναψη μιας συμφωνίας και το τι θα χρησιμοποιήσουμε από εκεί και πέρα για να συνομιλήσουμε και να συνεργαστούμε με μια χώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Madam Keller, Κύριε Κέλλα. Όλοι συμφωνούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικά και είναι σημαντικά όχι μόνο για τον ε, εξωτερικό κόσμο αλλά και για τις πολιτικές που εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ε, νομίζω ότι εκείνο που λείπει είναι να υπάρχουν τα σωστά εργαλεία για να μπορούμε να ελέγξουμε αυτήν την ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο είναι η αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει γίνει μερικέ φορέ, αλλά όχι για τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη αξιολόγηση επιπτώσεων για την ε, ε, Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών ή τη Συμφωνία Αλία ή την κοινή γεωργική πολιτική που τη μεταρρυθμίζουμε. Γιατί και εκεί, παραδείγματο χάρη, δεν εξετάζουμε τι επιπτώσει αυτή τη πολιτική στι ε, αναπτυσσόμενε χώρε. Η αξιολόγηση επιπτώσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι ερευνά κανείς ε, τις επιπτώσεις ε, που έχουν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες και όχι μόνο. Και αν γίνεται κάτι τέτοιο πιο συχνά μπορούν να έρθουν στο φως πολλές εμπορικές συμφωνίες που δεν βοηθάνε τελικά τους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι τους βοηθάνε τους εργαζόμενους αν θέλετε, τους εργάτες, απλούς εργάτες. Ένα άλλο εργαλείο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ είναι ένας μηχανισμός ε, διαμαρτυρίας ε, παραπώνων όπως ένα ομπουτσμαν όπου μπορούν να καταφύγουν οι άνθρωποι για να παραπονηθούν όταν ε, θεωρούν ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίω μπορεί κανείς να καταφύγει στις ΜΚΟ, αυτές απευθύνονται στις ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες συνεργάζονται. Δεν υπάρχει όμως θεσμοθετημένος οργανισμός ε, κατάθεσης παραπώνων. Πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλονται επίσης στην ασυνέπεια που υπάρχει. Ε, Παραδείγματος χάρη ε, η Συμφωνία Αλίας όπου αφαιρούμε έσοδα και ε, τρόφιμα από τους ανθρώπους του τρίτου κόσμου. Πρέπει λοιπόν εκεί να εφαρμοστούν οι σωστοί μηχανισμοί ε, και νομίζω αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατη αλλά νομίζω και στα κοινοβούλια. Κάτι τέτοιο ε, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας ως βουλευτές. <clears throat> Δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταθέτουμε ε, ε, ψήφισμα, εμείς ε, έχουμε έναν μόνιμο εισηγητή για την ανάπτυξη, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Και δεν πρέπει να περιμένουμε άλλους να εφαρμόσουν αυτά που πιστεύουμε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να στρέψουμε πιο προσεκτικά το βλέμμα το τι υπάρχει στα δικά σας κοινοβούλια, τι υπάρχει στα δικά μας, να εφαρμόσουμε καλύτερα μηχανισμούς και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε όχι απλά με πανηγυρικούς λόγους σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι να δούμε πώς μπορούμε να τα ε, εφαρμόσουμε στην πράξη. Ευχαριστώ και τώρα βλέπω ότι ζητούν και άλλοι το λόγο για να συμβάλλουν στη συζήτηση ή μήπω όχι. Δεν θέλω φυσικά να σας πιέσω, ίσως να έχουμε καλύψει και τα πιο σημαντικά ζητήματα. Δεν χρειάζεται οι πολιτικοί να μιλούν μόνο για να μιλούν. Εγώ νομίζω τουλάχιστον έμαθα πολλά στην συνάντηση αυτή, της συνεδρίαση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ήδη ότι εδώ στο Κοινοβούλιο θα αναλύσουμε σε βάθος την αιρεσιμότητα αυτή όταν περάσουμε στην εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά και την αναθεώρηση των μέσων για τα ανθρώπινα εργαλεία, για την ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα παραδόγματα τα οποία μας ε, δώσατε και υποθέτω ότι μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης θα γίνει μια αξιολόγηση της συνεδρίασης αυτής. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα συνεχίσουμε υπό την παρούσα σύνθεση. Εγώ για πρώτη φορά συμμετείχα και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επωφελής και χρήσιμη καρποφόρα πραγματικά η συνεδρίαση. Ελπίζω και εσείς να αποκομίσετε πολλά ωφέλη από την αλλαγή απόψεων και σας εύχομαι σε όσους έχουν έλθει εκτός Βρυξελών. Καλή επιστροφή στις πατρίδες σας. Σας ευχαριστώ.